εντελώς παράλογη συμφωνία γιατί για να αποφυφθούν οι ευρωεκλογέ, γιατί δεν θέλετε βέβαια να γίνουν, γιατί αν γίνουν θα κερδίσει το κόμμα του κύριου Φάραντς. Και αλλιώ αν δεν γίνουν αυτές οι ευρωεκλογέ στον Ηνωμένο Βασίλειο, επόμενες γενικές εκλογές εκεί θα κερδιθούν από το κόμμα του Brexit του κύριου Φάραντς. Οπότε λοιπόν αυτή η ευρωλατρεία πρέπει να φύγει από το Westminster. Ο κύριος Μπαρνιέ δεν είναι εδώ, ε. Πολύ καλός διαπραγματευτής. Και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, τη έκπληξή του, δεν θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιτυχία και λέει ότι δεν τη θέλει αυτή τη συμφωνία. Όμως, αυτή η ευρωολατρία είναι ακόμα πιο σημαντική για αυτούς που πιστεύουν ε, σε αυτήν και θεωρούν πιο σημαντικό να συνεχιστεί το οικοδόμημα αυτό όπως πηγαίνει τώρα, αντί να πετύχουν μια καλή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγείται με συνένεση και όχι με να θέλουν να τιμωρούν τους δε εκείνες τις χώρες, εκείνα τα άτομα τα οποία δεν συμμερίζονται την ίδια ευρωλατρεία. Συνεπώς, κυρίω από τι κάτω χώρε, ο κύριο Λάμπερτ, πρέπει ναι, να μαθαίνουμε από την ιστορία πράγματι αυτοί που έχουν ελεύθερη σκέψη από τις κάτω χώρε πρέπει να είναι παράδειγμα για μας. Δεν πρέπει να σταματάμε τον κόσμο από το να σκέφτεται και να αποφασίζει για τον εαυτό του. Η... Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η ιερά στην Ισπανία που οδήγησε. Αυτοί λοιπόν που σκέφτονται ελεύθερα σήμερα είναι αυτοί που εσείς ονομάζετε λαϊκιστές. Εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι λαϊκιστής παρά όχι μη λαϊκιστής όπως είσαστε εσείς. Αυτό που εσείς περιγράφετε ως λαϊκιστές πολύ σύντομα θα εκλεγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα έρθουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κυριαρχήσουν εδώ. Και θα αλλάξουν ριζικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα καταστραφεί αυτή. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να έχετε στο νου σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη απειλή στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, όπως ήταν η Ιερά Εξέταση τον 16ο αιώνα, που δεν επέτρεπε τη δημοκρατία και την ελεύθερη σκέψη. Κύριε, ο, ο Πρωθυπουργός Κάρενς είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τη μετανάστευση και ότι πολλοί θέλουν να έρθουν σε μια σταθερή δημοκρατική ήπειρο. Ε, δεν τους κατηγορώ. Κι εγώ, αν ζούσα στον τρίτο κόσμο ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ναι, κι εγώ θα ήθελα να έρθω εδώ. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, αλλά αν αλλάξουν τα νούμερα και αλλάξουν την ε, ίδια τη δημοκρατική φύση της Ευρωπαϊκής Υπήρου, τότε δεν ξέρω ποιοι θα θέλουν να πρωτοφύγουν από εδώ. Θα είναι μια καταστροφή. Το άλλο, ναι, είναι πιο ανησυχητικό από τα θέματα της υπηρεσίας υγείας. Τώρα, η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει μόνο αν κυβερνάται με συνένεση και όχι σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, έχετε δίκιο. Ο κύριος Κόμπουρν ξεπέρασε το χρόνο που είχε προβλεφθεί για εκείνον, αλλά άφησα και άλλους θα υπερβούν το χρόνο του. Ε, δεν είναι ότι όποιον συμπαθώ του δίνω χρόνο και όποιον δεν συμπαθώ δεν του δίνω. Οι κανόνε είναι όλοι για ίδιου. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Μπέι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, η τρομερή πυρκαγιά που χτύπησε την Παναγία των Παρισίων ε, μα κάνει να τη συνειδητοποιήσουμε το πόσο έφερε στο χαρακτήρα έχει η πολιτιστική μα κληρονομιά μα, να ένα από τα πιο ωραία κοσμήματα του ευρωπαϊκού μα πολιτισμού καταστράφηκε από τι φλόγε και μαύρησε την καρδιά των Γάλλων και των Ευρωπαίων. Ευτυχώ ε, η αξιοσημείωτη δράση των πυροσβεστών επέτρεψε να σωθεί ένα μεγάλο μέρο του κτηρίου που θα μπορέσει να αποκατασταθεί και να ξαναβρει το μεγαλείο του και με τη χαρά μαθαίνουμε ότι η θησαυρή τη ε, της των ε, Παρισίων ε, σώθηκαν ε, όπως τον Καθήνο Στεφάνη. Όμως όλο αυτό οδήγησε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κληρονομιά μας, αλλά και πιο γενικά την κληρονομιά του ευρωπαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερθήκατε προλίγο σε αυτό που αποκαλείται ευρωσκεπτικιστές και θεωρείτε ότι είναι αντίθετοι στην ίδια τη ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εδώ κάνετε 100% λάθος. Πιστεύουμε στην Ευρώπη, είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός, ένας κοινό πολιτισμός και υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Όμως αυτή η βούληση απαιτεί επίσης και διάβια πνεύματος. Και είπατε για τη μετανάστευση δεν έχω λύση, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε για να εμποδίσουμε τη μετανάστευση. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε να δράσουμε και το δείχνει καθημερινά ο Ματέο Σελβίνη στην Ιταλία. Όμω υπάρχουν δύο επιλογέ ξεκάθαρα. Αφενό, ο κύριο Αβραμόπουλο, ο Ευρωπαίο Επίτροπο, μα είπε ότι χρειαζόταν μετανάστευση για να καλύψουμε το δημογραφικό έλλειμμα. Και αφετέρου, η θεραλέα κυβέρνηση στην Ιταλία αλλά και στην Ουγγαρία που θεσπίζουν μεγάλε κοινωνικέ φορολογικέ πολιτικέ που υποστηρίζουν την οικογένεια και την ευρωπαϊκή γεννητικότητα. Υπάρχουν λοιπόν δύο οράματα εδώ που συγκρέονται μεταξύ αυτών που δέχονται και ενθαρρύνουν τη μετανάστευση και όσοι το αντίθετο θέλουν ε, να σταματήσει το μεταναστευτικό ρεύμα και να ενθαρρύνουν την ε, γεννητικότητα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από κατάργηση κάθε προστασία ε, με την εσωτερική αγορά, τον θεμητό ανταγωνισμό, με του απεσπασμένου εργαζομένου ε, και στο εξωτερικό, πολλαπλασιάζοντα ε, τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και τη μείωση των δασμών. Σήμερα, οι ΕΠΑ και η Κίνα προστατεύουν τον εαυτό του, μπορούν να προστατεύσουν με κάθε τρόπο την εσωτερική του αγορά και φυσικά έχουν επιθετική στάση στον υπόλοιπο κόσμο και χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ως ένα χώρο που μπορούν να δράσουν ελεύθερα, συνήθως ε, εις βάρος ε, της δικής μας οικονομίας και των εργαζομένων μας. Ορίστε και εδώ έρχονται ε, σε αντίθεση δύο οικονομικά οράματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ως ένα εντελώς ανοιχτό χώρο και ένα άλλο όραμα που να προστατεύεται οικονομικά και εμπορικά σε ό,τι αφορά τη θεσμική οργάνωση. Η Ευρώπη θα πρέπει ε, να προωθήσει την δημοκρατία μπροστά στην ε, τεράστια εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, άκουσα τι είπε και ο κύριος Βέμπερ και ο Μανώλ Μακρόν μας είπαν ότι πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά στο φεντεραλισμό και να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας. Επίσης μας ζητούν και να καταργηθεί και η δική η πλειοψηφία και τέλος και απλή πλειοψηφία για να καταλήξουμε σε μια εντελώς πιο αδιαφανή λειτουργία και πιο αυτα αυταρχική. Και εδώ έχουμε δύο αντιτιθέμενα οράματα, η Ευρώπη τη συνεργασία και των εθνών ή η Ευρώπη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιτάχυνση προ το φεντεραλισμό. Ε, απέχουμε πέντε εβδομάδες από τις ευρωεκλογέ. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, φυσικά είναι στο σταυροδρόμι ε, και έχει την ικανότητα η Ευρώπη να δώσει μια ευκαιρία προκειμένου να λάμψουν τα έθνη μας στην παγκόσμια σκηνή. Όμως θα πρέπει να σπάσουμε το μεγάλο δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και να απομακρυνθούμε από τη τεχνοκρατική λογική. Η Ευρώπη θα προστατεύσει την οικονομία της ή θα γίνει ο εξυπηρέτηση των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Η Ευρώπη θα θέσει τα έθνη και τους λαούς ε, στο κέντρο του προγραμματός της ή θα διαλυθεί, θα υπερασπίσει τον πολιτισμό της ή την ταυτότητά της ή θα εξαφανιστεί. Ο κύριος Γκόλνης από τους μια εγγεγραμμένους, παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ και αγαπητέ τελευταίο συνάδελφε, μας μιλάτε για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν φαίνεται αυτό το μέλλον πολύ λαμπρό αν δεν αλλάξουμε προπτική. Τα 30 χρόνια που είμαι εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα να αναπτύσσεται μια στρεβλή δυναμική των πολιτικών ομάδων ε, που θυμίζει κακές στιγμές. Πρόκειται για τις αρχές που διακηρύσει χωρίς όμως να τηρεί και έτσι είναι σε βάρος των διαφόρων μειονοτήτων. Νομίζουμε ότι έχουμε εντολή για να κανονίσουμε τα πάντα, ακόμα και τη σεξουαλική ζωή των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα υπερκράτος παγκόσμιο που να έχει ένα σωρό περιορισμούς κανόνες, αλλά να είναι ανοιχτό σε ανταγωνισμό με χώρες που δεν έχουν τίποτα ή πάρα πολύ λίγα. Η δικιά σας χώρα απελευθερώθηκε από το ζυγό της ε, σοσιαλιστικής χώρας ε, στην οποία βρισκόσαστε. Δεν νομίζω ότι θέλετε να έρθετε εδώ για να βρεθείτε σε έναν άλλο ζυγό. Πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές αξίες του πολιτισμού μας. Να υποδέχεται τη ζωή και όχι την άμβλωση τη μαζική. Να θέλει την οικογένεια και όχι να την καταπιέζει συστηματικά όπως επίσης τις ε, σεξουαλικές μειονότητες. Εμπόρια, ε, πορικά αγαθά. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που προσφέρει την ευτυχία και την ευημερία. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ ελεύθερων εθνών με συγκεκριμένα προγράμματα, με νούμερα και σε συγκεκριμένους τομείς όπου ο πολίτης να μπορεί να μετρήσει και το κόστος αλλά και το ωφέλη. Η επανάσταση των λαών κατά εκείνων που θέλουν να τους περιορίσουν, που περιορίζουν την ταυτότητά τους, έχει ξεκινήσει. Και εδώ ακόμα καταφέραμε να ρίξουμε τα τείχη του ψεύδους που εμπόδιζαν τους πατριώτες από διάφορες χώρες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε αυτό λοιπόν το βελούδινο περιβάλλον υποκρισίας οι λαοί αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια τους. Έχουμε σπήρι, άλλοι θα μαζέψουν τη συγκομιδή και για να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μας πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ζήτω οι ελεύθεροι λαοί μέσα σε μια ανανεωμένη Ευρώπη των Εθνών. Πρόεδρος, ε, ήμουνα ευέλικτος ε, στον πρώτο γύρο των παρεμβάσεων, αλλά επειδή στις 12.30 πρέπει να ψηφίσουμε και θέλουν να μιλήσουν όλοι εκείνοι ε, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία Catch the Eyes, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο που σας έχει δοθεί, γιατί αλλιώ θα αποκλείσετε κάποιους από το να λάβουν το λόγο. Και επειδή αυτή είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να φύγουν όλοι από την ολομέλεια ικανοποιημένη. Συμπεριλαμβανομένου και του Λετωνού Πρωθυπουργού, του κυρίου Κάρενς. Έχετε το λόγο για να δώσετε τις απαντήσεις σε αυτό τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μου παρέμβαση ήταν λιγάκι μακρά. Αυτή η παρέμβασή μου θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίζει κανείς τις διαφορές απόψεων. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή συζήτηση, ακούει ένα την άποψη του άλλου, σέβεται τον άλλον και τελικά ε, γίνεται η ψηφοφορία και προχωράει κανείς παρακάτω. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ε, για να γίνονται τα πράγματα, κάτι που η δική μου χώρα το βίωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν ήταν υπό την κατοχή της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή να μην έχει κανείς το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, να μην λέει τίποτα, κάποιος άλλος λαμβάνει τις αποφάσεις και σε συμπαρασύρει ή σε αφήνει κατά μέρο καθώς ε, προχωράει. Ε, νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές ε, ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος ανάμεσα στους δύο. Εγώ είμαι πρόθυμος ε, να συνεργαστώ με όλους όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Αυτή είναι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός καθώ να διατηρήσουμε νομιζω οτι ειναι απολυτα σαφες ποιο ειναι ο καλύτερο τροπος αναμεσα στου δυο εγω ειμαι προθυμος να συνεργαστω με ολους οσοι πιστευουν οτι πρεπει να προχωρησουμε μαζι αυτη ειναι η δυναμη της ευρωπαικης ενωσης το γεγονό οτι κατορθωσαμε να διατηρησουμε ε κυριαρχες χωρες με ισχυρες ταυτότητες με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους η κάθε μία, με ιστορία που βέβαια συνδέεται μεταξύ των διαφόρων χωρών πολλές φορές και παράλληλα κατορθώσαμε να ανοίξουμε τις αγορές στο εμπόριο. Μπορέσαμε να συνδυάσουμε, να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και να εκφράζουμε μια ισχυρή φωνή στον κόσμο. Για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι η Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Μα απολύτως τίποτα. Εδώ έχουμε μία ένωση ελεύθερης πολιτικής βούλησης. Ε, τα κρατημέλη είναι ελεύθερα να συμμετέχουν, οι πολίτες επίσης ελεύθεροι να συμμετέχουν και βλέπουμε ότι αν οι πολίτες αλλάξουν γνώμη, κανείς δεν τους εμποδίζει. Είναι μια πραγματικά ελεύθερη ένωση, είναι ένα μοναδικό εγχείρημα στον κόσμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια χώρα που βασίζεται προέκυψε από τη μετανάστευση. Οι αρχαίγονοι Αμερικανοί δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχουν πολλοί εξ αυτών. Αυτοί τους οποίους ε, αποκαλούμε Αμερικανούς ε, σε γενικές γραμμές έρχονται από την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Ε, αφήνουν κάτι πίσω τους και γίνονται κάτι καινούριο όλοι μαζί. Στην Ευρώπη όμως κανείς από εμά δεν είναι αναγκασμένος να μετακινηθεί. Μπορούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, την ταυτότητά μας και συνεργαζόμαστε σε πολιτικό και οικονομικό πεδίο για να εκφράσουμε τα κυρίαρχα συμφέροντά μας. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν παρετούμεθα από τίποτα, συνδυάζουμε τους πόρου μα και από το να είμαστε απομονωμένοι και μεμονωμένοι είμαστε πολύ πιο ισχυροί ως μια ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Πρωθυπουργέ για την σύντομη ομιλία σας. Ο πρώτος που έχει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ είναι ο κύριος Κέλαμ. Κύριε Πρόεδρε, και για μένα αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα νομίζω όσον αφορά την ρωσική επιθετικότητα πρέπει να διερωτηθούμε τι μπορεί να γίνει ακόμα και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει στο να εξισωθούν τα ε, εγκλήματα των ε, κομμουνιστών με αυτά των Ναζί. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει. Εάν η ΚΑΓΚΕΜΠΕ της ε, Σοβιετικής Ένωσης ε, όπως και η Γκεστάπο του Χίτλερ είχε καταδικαστεί με τον ίδιο τρόπο ως δολοφονική οργάνωση, τότε και τα στελέχη της Γκεστάπο, της Γκεστάπο, της Καγκεμπέ δηλαδή, της Ρωσίας, δεν θα μπορούσαν ε, σήμερα να ηγούνται της Σοβιετικής Ένωσης. Το κράτος που υπάρχει σήμερα υπάρχει μόνο λόγω της ε, διαφθοράς, της ευρωπαϊκής διαφοράς, ε, κλάπησαν χρήματα και οι Ρώσοι τα ξέπλυναν σε δυτικές τράπεζες. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτές τις ροές χρημάτων, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πλέον, δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο κύριος Πούτιν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλαμ που για τόσα χρόνια ήταν υποδειγματικό βουλευτή. και το έχω πει δημόσια. Για μένα πάντοτε αποτελούσατε παράδειγμα προ μίμηση. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση και θαυμασμό για σας, ε, γιατί έχετε αγωνιστεί για την ελευθερία της ε, χώρας σας και για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συνεισφορά στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόπες Αγγιλάρη είναι ο επόμενο ομιλητή, Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κύριε Πρωθυπουργέ. Πρόκειται για το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να δείξουμε σεβασμό στο είναι ομιλία σας υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, είναι καιρό να αποτιμήσουμε τις συζητήσεις που είχαμε με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Να χαιρετήσουμε το έργο του Προέδρου Γιούνκερ ο οποίος έδωσε υψηλής ποιότητας απαντήσεις. Όμως, θέλω να πω κάτι αφού άκουσα την ομιλία σας. Μιλήσατε ε, όχι για την καταπολέμηση του λαϊκισμού, αλλά δεν είναι ασυμβιβαστό να τον καταπολεμήσουμε όταν ακούμε τέτοιες ε, ανοησίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να απαντήσουμε. Δεύτερον, μιλήσατε για τη μετανάστευση. Ναι, πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είπατε τίποτα για αλληλεγγύη. Και αυτό αποτελεί μια εντολή τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και ε, την διαχείριση των συνόρων, ε, τότε αυτά θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ Κάριν. Σταρμπάτη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Jean-Claude Juncker είπε ότι πρέπει κανείς να αγαπάει την Ευρώπη. Δίκιο έχει, και εγώ την αγαπάω. Αλλά ακριβώ όταν αγαπάει κανείς την Ευρώπη πρέπει να κατανοεί και τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέω ότι δεν πρέπει να θυσιάσουμε τους λαούς μας στο βωμό της Ευρώπης Κύριε Ντομπρόφσκι, ε, ε, ξέρετε ότι οι νέοι μας ε, φεύγουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην μεταναστεύουν. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς είπατε ότι ε, χρειαζόμαστε αγορές μη ρυθμισμένες και έχουμε δύο κεντρικές αγορές που είναι απόλυτα ρυθμισμένες και έχουμε τις ισοτιμίες και τα επιτόκια. Εάν λοιπόν είναι συνεδεμένες οι ισοτιμίες με τα επιτόκια, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να παρισφρήσουν άλλοι παράγοντες, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, τότε υπάρχει ένας σκληρός μηχανισμός προσαρμογής στην αγορά. Εύχομαι λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο μέλλον, να μην λέει κανείς ότι ε, πρέπει να θυσιάσουμε τους λαούς μας στο βωμό της Ευρώπης. Όχι. Το εργατικό δυναμικό πρέπει να υπάρχει εδώ στην Ευρώπη. Το να ε, μην φροντίζουμε τον ανταγωνισμό, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα κράτη πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να επιτελέσετε στο μέλλον. Ο κύριος Πιτροφάνο, τους παρακαλώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικά Ήθελα να μιλήσω για την φυγή εγκεφάλων ε, που βιώνουμε στη χώρα μας, ε, τη Λετωνία. Εμείς ε, χάνουμε τους νέους ερευνητέ μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να αντιδράσω σε ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Γιατί ζήτησε από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα τη ολοκλήρωση στη Λετωνία. Πρέπει να πω, δεν είναι μια ιστορία επιτυχία. Είναι μια ντροπιαστική ιστορία ε, που στρέφεται κατά τη εκπαίδευση των μειονοτήτων. Ε, μετά την ανεξαρτησία, το μεγαλύτερο μέρο των μειονοτήτων ε, υποστήριζαν ε, την ανεξαρτησία και την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης χώρας. Όμως ε, τώρα τα παιδιά μας, δεν, τα παιδιά των οικογενειών των μειονοτήτων δεν μπορούν να μορφώνονται στη μητρική τους γλώσσα. Παρακαλώ μην ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα συνάδελφοι. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για 2.000 χρόνια στην χώρα μου είχαμε αυτή την τρέλα για την Ευρώπη. Η δικιά μου η χώρα δεν είναι ευχαριστημένη με την Ευρώπη. Όταν έχεις σωθεί από τα πεδία των μαχών, εξακολουθείς και θέλεις να πιστεύεις, θέλεις την ειρήνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό ήταν ένα πείμα ενός Ούγγρου ποιητή το 83 και εσείς ε, ακούσατε τα πρώτα και τα τελευταία λόγια του πείματος αυτού. Και αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Θεός να φυλάει και να προστατεύει τη χώρα μου και τη χριστιανική Ευρώπη. Αντίο σας. Ο κύριος Βέρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Λετωνίας, σας θαυμάζω πολύ, όχι μόνο γιατί γίνατε Πρωθυπουργό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε αναλάβει αυτό το καθήκον. Ήσασταν και προβλεφτή τώρα είσαστε από ένα μικρό κόμμα, καταφέρατε όμως να πετύχετε πλειοψηφία και να ηγηθείτε επιτυχώς τη σημερινή κυβέρνηση στη Λετωνία. Πράγματι, αξίζετε γι' αυτό, γιατί είσαστε ειλικρινής, τίμιος και έχετε πάρα πολλές ικανότητες. Είσαστε μια επιτυχής ιστορία. Αυτό είναι και η ιστορία της Λετωνίας. Βέβαια, τώρα η βασική ερώτηση. Ζείτε σε μια χώρα που βρίσκεται σε μετάβαση, όπω και η δικιά μου η Σλοβενία. Το θέμα του κράτου δικαίου είναι πάντα πολύ επίκαιρο. Ήμασταν μάρτυρε ε, των ε, διαφόρων ε, κομμάτων και παραδόσεων και επεισοδίων που παρακολουθούμε. Εγώ πιστεύω ότι και άλλες χώρες σε μετάβαση έχουν προβλήματα με την δικαστική εξουσία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχει δηλαδή έναν μηχανισμό ώστε όταν υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου σε χώρες μετάβαση να κάνουν κάτι. Ευχαριστώ, η κυρία Πιλάρντε Καστιγιώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχουμε μπροστά μας ε, τον Πρωθυπουργό, είναι ένας εξαιρετικός ε, συνάδελφος, αλλά ε, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κάρνης. Θέλω να πω ότι αφήσατε το αποτύπωμά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι τότε που ήσασταν συντονιστής, που είχατε υπό την καθοδήγησή σας πολλά σημαντικά θέματα. Αυτό όμως που σήμερα είναι το πιο σημαντικό είναι ότι μας παρουσιάσατε ένα όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για το παρελθόν, το παρόν και το πιο σημαντικό για το μέλλον. Και ε, σε αυτό τον δρόμο πολύ σωστά αναφέρατε και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η κοινή αγορά. Πιο συγκεκριμένα η ενιαία ψηφιακή αγορά. Αναφέρατε το που ακριβώς βρισκόμαστε και ξέρετε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο διστάζει. Δεν είναι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο δεν αναχαιτίζει τους φραγμούς. Τώρα εσείς έχετε μία ε, πλεονεκτική προνομιούχο θέση στο Συμβούλιο, έχετε έντρα, Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έτσι μπορείτε να προχωρήσετε πολύ πιο γρήγορα και να άρετε τους φραγμούς. Σας εύχομαι καλή τύχη. Καμπούλα Νάτρη, επόμενη ομιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή να γνωρίζω τον Πρωθυπουργό ως καλό συνάδελφο στην Επιτροπή Ήτρε τότε που εργαζόμασταν για μια ε, ψηφιακή ενωμένη Ευρώπη. Ε, πραγματικά και εγώ με πολύ χαρά εργάζομαι για αυτήν την Ευρώπη όπου θα είμαστε αρκετά θαραλέοι για να εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι μπορούμε μόνο από κοινού να, παρουσιά, να επιτύχουμε πάνω από 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ε, άρα λοιπόν αυτό το 20% είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα λαϊκίστικα που αναφέρονται, κλείστε τα σύνορα ή ε, μην κάνετε εμπόριο με άλλες περιοχές, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πώς αυτό θα βοηθούσε τους Ευρωπαίους. Αλλά όταν μιλάμε και για την κλιματική αλλαγή και εκεί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι από κοινού μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, απλές οικογένειες που θέλουν να έχουν αυτοκίνητο. Όμως η αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει νέα αυτοκίνητα με μικρότερες ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε όλοι από κοινού. Ως εκ τούτου προσβλέπω στο να απευθυνθεί η Ευρώπη στους ε, πολίτες της και κατά διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία. Νομίζω όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι εμείς έχουμε δουλέψει για να μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινούνται και πέρα από τα σύνορα, δουλέψαμε για να υπάρχουν καλύτερε συνθήκε εμπορίου και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ντεσμέικερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάριν. Πολύ ισχυρή η ομιλία σας, πολύ δυνατή για τα δημοκρατικά έθνη. Ωραία. Small is beautiful. Και η Λετωνία είχε κυριαρχία από πολύ ισχυρού γείτονε για πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχει καταφέρει να έχει μια τεράστια επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπει αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλα έθνη, η Σκοτία, η Καταλωνία, που είναι ε, δημοκρατικά και δημοκρατικά προσπαθούν να ανεξαρτοποιηθούν και όμως αυτό φαίνεται να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ. Και εξού και η βία σε βάρος των ψηφοφόρων στην Καταλωνία από τους ηγέτες της Ισπανίας. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μόνο όταν δούμε ότι το δημοκρατικό δικαιώμα, τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών γίνονται σεβαστά. Και δεν μπορεί να μιλάμε χωρίς να κάνουμε αυτά που λέμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Οι εξελίξεις στην Λετωνία, την Εστονία, τη Λιθουανία αποτελούν το θαύμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Καταπληκτικά επιτεύγματα. Ελευθερία. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα στην Σουηδία να στηρίζω. Ε, πριν στήριζα την ανεξαρτησία της Εστονίας, της Λετωνίας, της Λεθονίας, θυμάμαι, με τη Σάντρα του και ένα σωρό άλλους. Αγωνιζόμασταν για την ανεξαρτησία στην Σοβιετική επικράτεια. Και τώρα ένας καλός μου φίλος, εδώ δίπλα μου κάθεται, και εσύ ναι, Ήτανε ευρωβουλευτής και τώρα είναι επικεφαλής της κυβέρνησης της ελεύθερης Λετωνίας. Αυτό είναι το θαύμα. Και θέλω να το πω σε όλους τους συναδέρφους εδώ, γιατί και για μένα αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ. Ωραία, θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να σας είχαμε εδώ, Κριστιανής Καρίνης. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω, δεν χρειαζόμαστε τους Φάρατζης και, και τους Κόμπερνς εδώ πέρα που να μας λένε ότι είναι καλύτερα να μην έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτά που εσείς καταφέρατε είναι ακριβώς ένα τεράστιο επίτευγμα. Μας δείξατε, είσαστε το ζωντανό παράδειγμα το ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και τι ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε. Εσείς, οι χώρα σας, οι χώρες μας είναι το καλύτερο παράδειγμα της Ευρώπης και είμαστε περήφανοι εμείς οι Σουηδοί, γιατί είμαστε από τη Σουηδία, που σας είχαμε και, τον, και σας έχουμε γειτονική χώρα. Ευχαριστώ, Γκούναρ, ε, για το έργο σου στο Κοινοβούλιο αυτό. Συνάδελφος Μπόγκοβιτς. Καλημέρα σας, αγαπητέ Γεστίαν. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να σε ξαναβλέπω. Είχαμε περάσει πολύ καλές στιγμές ως συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σου. Σλοβένος Σλοβαίνος Πρωθυπουργός ε, είχε ε, προσκληθεί να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως απέριψε την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ λοιπόν για την υπέροχη ομιλία σου που ολοκληρώνει αυτό το ε, επεισόδιο όταν έρχονται οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να μιλήσουν για το μέλλον της Ευρώπης. Η χώρα σου είχε μία δύσκολη ιστορία αλλά και εσύ είχες πέρα μια ιστορία, προέρχεσαι από μετανάστες γονείς και θαυμάζω τώρα πόσο δεσμευμένος είσαι για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αφενός και πόσο αφοσιωμένος είσαι στην ελευθερία αφετέρου. Είπες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και σε ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας, στην οικονομία κτλ. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέλω να θέσω την εξή ε, ερώτηση. Οι καθαροί συνεισφέροντες στο Συμβούλιο κατανοούν ε, ε, την έννοια της ελληνικής που μπορεί να εκφραστεί μέσω της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής αξίζει για να ε, καταβάλουν το 1 τρίτο, συγγνώμη, το 1,3 του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Εγώ ελπίζω όμως ότι θα γίνει η Ευρώπη καλύτερη στο μέλλον. Μπλάνκο Λόπε, παρακαλώ, που είναι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Τη διάρκεια αυτή της θητεία ε, μπορέσαμε να συνεργαστούμε και το λέω στην τελευταία μου παρέμβαση αυτό στο Κοινοβούλιο. Να συνεργαστούμε λοιπόν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πιο ανταγωνιστική, με λιγότερες εκπομπές άνθρακα μαζί και με τον Επίτροπο Κανιέτα για να συνεργαστούμε για να έχουμε μια νομοθεσία που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι η μεγάλη απειλή κατά του πλανήτη έχοντας μια οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα ιδιαίτερα φιλόδοξη. Γιατί ξέρουμε ότι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται είναι η πιο καθαρή. Να συνεργαστούμε για την οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση και σίγουρα μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών του άνθρακα σε τομεί που ρηπαίνουν όπω. Ε, είναι η θέρμανση, η ψήξη και οι μεταφορές. Να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τις εκπομπές και για να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καθολικό νομοθετικό πλαίσιο που να μας καθιστά ε, σε μια ηγετική θέση για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει μέλλον να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όπως πράξαμε σε αυτή τη θητεία καταπλημώντας το είναι πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ για τη δική σας συνεισφορά. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα ακούσαμε επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο παρουσιάζουν ε, εντυπωσιακά νούμερα και αναφέρετε και παραδείγματα. Συνεργαστήκαμε για θέματα καταπολέμησης της ε, διαφθοράς, επίσης ε, για την αντιμετώπιση της, παράνομης, της νομιμοποίησης από παράνομα έσοδα όσον αφορά αυτό το ξέπλυμα του χρήματος δεν είναι μόνο τα χρήματα που έρχονται από εγκληματικέ δραστηριότητε, αλλά και τα χρήματα που διοχετεύονται στην τρομοκρατία, στην παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων. Στο επόμενο λοιπόν κοινοβούλιο θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εκτενώς ε, για τα θέματα αυτά. Επόμενος ομιλητής, Βαϊτέρε, παρακαλώ, η κυρία Βαϊτέρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Πρωθυπουργό μας. Ε, η ομιλία σου ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ανέφερες και πολλά επώδυνα θέματα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Είμαι επίση ε, ιδιαίτερα υπερήφανο ε, που κατόρθωσε ε, να συστήσει κυβέρνηση στην Λετωνία και με νέε δυνάμει όταν ε, παλιά στελέχη φοβόντουσαν. Εσύ όμως τα κατάφερες, μπροστά μας ε, έχουμε πολλά και δύσκολα. Βεβαίως ε, πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες μας, διότι δεχόμεθα πλέον λιγότερα κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άμεσες ε, πληρωμές ε, είναι μικρότερες από ό,τι σε άλλες χώρες ε, και όσον αφορά την κοινωνία ακούσαμε ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική ρωσοποίησης και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε κατά αυτής. Αναφέρθηκαν και τα θέματα μειονοτήτων. Η Λετωνία είναι η μόνη χώρα όπου εξακολουθούμε να προσφέρουμε μια πλήρη ρωσική εκπαίδευση γλώσσα μιας ε, χώρας ε, μπορεί να πίσταται διακρίσεις. Δύσκολα όλα αυτά για τη Λετωνία, αλλά ε, στο μυαλό μας είναι η ασφαλής Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σας εύχομαι καλή τύχη. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας η οποία ήταν ρεαλιστική και εύρωστη αλλά και για τις ρεαλιστικές και συνεκτικές αξιολογήσεις και συνεισφορές σας. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε. Και εγώ και η χώρα μου, η Ρουμανία, βλέπουμε την Ρωσία όπως τη βλέπετε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, πώς η Λετωνία αξιολόγησε την, αξιολογεί την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και ποια θα πρέπει να είναι μελλοντική σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σας ευχαριστώ. Μπένσεν. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που παρουσιάζετε ένα όραμα εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις σας για την εσωτερική αγορά θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο, να πείτε ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα απειλούνται από την κομμουνιστική Κίνα. Αυτό που έχουμε τώρα ενωπιών μας και βλέπουμε είναι η βιομηχανία των ευρωπαϊκών πλοίων που δέχονται επίθεση από τον κινέζικο ανταγωνισμό. Ε, βλέπουμε κάποια ναυπηγεία που πρέπει να πάρουν επιδοτήσεις ε, για να παροπλήσουν ε, τα παλιά πλοία τους και κατόπιν θα πρέπει ε, να προσαρμοστούν στις απαιτήσει των κινέζικων εταιριών για την αυπήγηση των πλοίων. Πρόκειται για θέμη του ανταγωνισμό απέναντι στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό αυτοκλάδο. Και βλέπουμε ότι κατακτούν μια αγορά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αγορά Ευρωπαίων ιδιωτών χωρίς να υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις. Όμως δεν θα πρέπει να είμαστε ανόητοι. Εδώ θα πρέπει η Κομισιό να τα σκεφτεί όλα αυτά πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο κύριος Ρανζέλ. Ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ κύριε Πρωθυπουργέ για μία από τις πιο εμπνευσμένες ομιλίες που έχουμε ακούσει εδώ από πρωθυπουργούς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την πολιτική συνοχής και τα ταμεία συνοχής. Η Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση μια χώρα όπως η Λετωνία που έχει καταβάλει τόσες προσπάθειες και βρίσκεται σε χαμηλή θέση του χαμηλού μεσόρου χάνει 14% από το Ταμείο Συνοχής. Η Πορτογαλία χάνει 7%. Η Κροατία χάνει 5%. Είναι αποδεκτό οι πιο φτωχές χώρες να χάνουν κονδύλια από την πολιτική συνοχής. Πώς ο Πρωθυπουργό Κάρνη σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, ε, θα δράσει όπως η Πορτογαλική κυβέρνηση, που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ικανοποιημένη, που η Κομισιόν από χώρε που είναι πιο φτωχέ, από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία και έχουν σεβαστεί όλη την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, να του αφαιρούνται κονδύλια από την πολιτική συνοχή. Ε, ποια μέτρα μπορούν και πρέπει να λάβουν οι χώρε αυτέ απέναντι στην πρόταση τη Κομισιόν. Ο κύριος Μίμικινς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, στην ομιλία σας δείξατε και το κινητό σας, μιλήσατε και για τον μύθο του Εσώπου. Οι διαφορές και η ποικιλομορφία στην Ευρώπη, ναι, υπάρχουν. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι έστειλαν επιστολή στην λετονική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εκπαίδευσης της γλώσσας των μενοτήτων τους αποκαλέσατε τρελούς. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία ε, Μάλλον είχατε και μια έκθεση πάρα πολύ καλή για το ξέπλυμα του χρήματος, αλλά δεν είπατε τίποτα για την ε, σύζυγό σας και για τις πωλήσει ακινήτων. Είπατε ότι είναι ο τύπος. Ναι, ίσως να μην είναι καλό ε, παράδειγμα. Αν θέλετε κύριε Κάνης να αλλάξετε την Ευρώπη, πρέπει να ξεκινήσετε από τον εαυτό σας. Δεν πρέπει να έχετε πια αμερικανική υπηκότητα. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάριντς. Θέλω να σας θυμίσω ένα πράγμα εγώ, κύριε Κάριντς. Πριν από 10 χρόνια θυμάμαι ότι πήγα στην ε, καντίνα και ήμουνα κάπως μόνος, γιατί και εσείς και κάποιοι συνάδελφοι με καλέσατε να έρθω και να μοιραστώ το γεύμα μου μαζί σας, να καθίσουμε μαζί. Δεν το ξεχνάω και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ και για αυτά που είπατε χτες στην συνεδρίαση της ομάδας του ΕΛΚΑ. Τώρα, αναφερθήκατε όντως στο ξέπλυμα χρήματος και στην εγκληματικότητα. Και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα στη χώρα σας και είπατε πώς ε, κυκλοφορούν εγκληματίες από τη μία χώρα στην άλλη. Εσείς τι θα θέλατε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία για να μειωθεί ακριβώς η νομοποίηση χρήματος από παράνομες ε, δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι σας καλωσορίζουμε εσάς και τους συναδέλφους σας εδώ. Η κυρία Γκόμες. Σας ε, καλωσορίζω κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και χάρηκα πάρα πολύ που συνεργαστήκα μαζί σας ε, στην ομάδα που διαπραγματεύτηκε την τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για το ξέπημα βρώμικου χρήματος. Όπως και εσείς και εγώ έμαθα πάρα πολλά και λόγω των ε, επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα και για θέματα φορολογικά. Εκτιμώ αυτά που είπατε και σας στηρίζω ανεπιφύλακτα ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή κεντρική εποπτεία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σας ερωτώ όμως, εσείς τώρα ως ε, Πρωθυπουργός θα πιέσετε και για αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς την πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Επίσης για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ ε, θα ασκήσετε εκεί πίεση γιατί βλέπουμε ότι διοχετεύονται πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα από το, τις απάτε απάτες ε, καρουσέλ. Και σας ερωτώ, θα πιέσετε για το MQV σε θέματα φορολογίας. Αυτό είναι καθοριστική σημασία ε, για να αντιμετωπιστεί κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φορολογικό dumping το οποίο στρεβλώνει τους, ε, αγώνες θεμητού, κανόνες θεμητού ανταγωνισμού. Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι πάρα πολύ που ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ε, βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ε, Πρόεδρε, αυτά που είπατε σήμερα ήταν ε, ρεαλιστικά, θετικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός σε όλα τα κράτη-μέλη, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Ο καλύτερο τρόπος είναι να καταδείξουμε ότι έχουμε ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι μόνο μόνο ένα εγχείρημα ειρήνης, αλλά είναι και ένα εγχείρημα οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου. Και το θεματολόγιο σας, Πρόεδρε, είναι σαφές. Θέλετε περισσότερο εμπόριο, να έρθουν οι φραγμοί που εμποδίζουν την κοινή αγορά, να μην υπάρχει προστατευτισμός, με περισσότερες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμητός ανταγωνισμός. Αυτό είναι το θεματολόγιο που θα διασφαλίσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, περισσότερες επενδύσεις, αλλά και περισσότερες ελπίδες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας. Σας στηρίζουμε και εκτιμούμε όλα αυτά που κάνατε για τη δημοκρατία, την ελευθερία, για τις αξίες για τις οποίες τόσο εύγλωτα μιλήσατε σήμερα το πρωί. Ο κύριος Βάιντεν Όρτσελ δεν είναι εδώ. Μερκούνεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε αντίθεση με άλλους συναδέρφους, ε, δεν είναι η τελευταία φορά που εγώ μιλάω εδώ στο ημικύκλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάριν, τον Πρωθυπουργό, για την ενέργειά του, για την τόσο θετική ομιλία του για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα να συνεργαστώ μαζί σας αυτά τα χρόνια. Η προτεραιότητα ήταν η δημιουργία απασχόλησης επενδύσεων και εταιριών. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Έχουμε περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη σήμερα, έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες επενδύσεις σε βαθμό όπως ήταν πριν από την κρίση. Όμω είναι δύσκολος ο διεθνή ανταγωνισμός, η ψηφιοποίηση αλλάζει τον κόσμο, οπότε εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνουν οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητά μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε κύριο Βαλσίτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την εξαιρετική ομιλία σας. Εσείς αναφερθήκατε στην ιστορία όχι μόνο της Λετωνίας, αλλά και των άλλων βαλτικών χωρών, της Εστονίας και της Λιθουανίας. Ε, δεν θέλω να σας κάνω ερωτήσεις, αλλά βλέπετε είναι η τελευταία μου ομιλία στο ημικύκλιο αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Και θέλω να κάνω έκκληση σε εσά, να σας ενθαρρύνω μια που είσαστε εκπρόσωπος του Συμβουλίου, να στηρίξετε την δημιουργία μιας αυθεντικής ενεργειακής αγοράς. Και δεύτερον, θέλω να κάνω έκκληση σε εσά να στηρίξετε επίσης και το πρόγραμμα για σιδηροδρόμους στην Βαλτική. Να επικεντρωθείτε επίσης σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και επίσης πολύ σωστά τίθεται και το θέμα των πληρωμών ε, γεωργικών κονδυλίων, κονδυλίων προς την γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κάραντς ε, γιατί στην ομιλία τον έφερε κάτι το πολύ σημαντικό, δηλαδή την ε, ψηφιακή εσωτερική αγορά. Και Κρίστιαν έχεις απόλυτα δίκιο ότι αν δεν ε, καταργήσουμε τους φραγμούς στην Ευρώπη, κυρίως την περιαγωγή, ποτέ δεν θα κατορθώσουμε αυτές τις πλατφόρμες που τους χρειαζόμαστε πηγών στην Ευρώπη, αυτές να είναι και αποτελεσματικές. Χρειαζόμαστε την δυνατότητα να μπορούμε να αγοράσουμε κάρτα SIM και στα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρειαζόμαστε ουσιαστικές εξελίξεις γιατί αυτές θα καθορίσουν τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που από κοινού εργάστηκαν για την κοινή αγορά και διασφαλίζουν τον μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σας ευχαριστώ για αυτή τη φανταστική ευκαιρία Αγαπητοί συνάδελφοι, για πολλούς εδώ είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν ε, να μιλήσουν για μένα είναι πρώτη και τελευταία, καθώ πρόκειται για μένα. Είμαι ένα πολύ νέο μέλο, μόλι πριν δέκα μέρε ε, ήλθα. Και έτσι λοιπόν για στατιστικούς λόγους μήπως μπορείτε να σημειώσετε ότι είναι η πρώτη και η τελευταία μου παρέμβαση. Σας ευχαριστώ όμως ε, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να θέσω την ίδια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ο Ρουμάνος συνάδελφος. Ποια είναι η άποψή σα για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η Ρωσία έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, κατέχει, έχει κατα... παράνομα ε, μέρη της Ουκρανίας, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό και πώς ε, βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η δύσκολη σχέση με τη Ρωσία και ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα έπρεπε να σας δώσω και ένα δεύτερο λεπτό, αλλά δυστυχώς ε, δεν γίνεται. Συνάδελφος Αντρικιένε είναι εδώ στην αίθουσα. Τότε ολοκληρώνεται το κατσιδιάι και θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό. Έχετε το λόγο, κυρία Κάρινς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ κρατούσα σημειώσεις ε, όσο μιλούσατε. Έχω πάρει πολλές σημειώσεις ε, και φυσικά θα τις μελετήσω στο εγγύς μέλλον τα θέματα. Συνοχή, γεωργία, μετανάστευση, νομιμοποίηση συνόδων, Κίνα, Ρωσία, άμυνα και τα λοιπά. Αν προσπαθούσα να απαντήσω, μάλλον θα μακρηγορούσα πολύ περισσότερο από ότι την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν δεν θα το πράξω. Αλλά τι θέλω να κάνω, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ως πρώην ε, Ευρωβουλευτής θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ευκαιρία, την ικανοποίηση και την τιμή που είχα να συνεργαστώ μαζί σας. Τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά και η προηγούμενη θητεία ήταν ε, μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Από ό,τι φαίνεται συγκινούμε και κάπως. Όμως ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ καλή συνεργασία. Πολλοί από εσά είπατε ότι πρόκειται για την τελευταία ομιλία σα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω Πρωθυπουργό. Είμαι πολύ ικανοποιημένο λοιπόν γι' αυτό για να συνοψίσω τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια, συνάδελφοι. Δεν είναι τέλεια. Και όταν οι ψηφοφόροι μας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ακούσουμε τους ψηφοφόρους. Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όλα είναι τέλεια. Πρέπει να τους ακούσουμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πραγματικέ ανησυχίε. είτε πρόκειται για τη δουλειά του, είτε πρόκειται για τη μετανάστευση, το κλίμα, την ασφάλεια. Αυτά τα θέματα είναι πραγματικά, αλλά επίσης έχουμε και πραγματικές απαντήσεις στα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να εργαστούμε στο μέλλον ως ε, μια ένωση ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών ε, χωρίς να ε, δίνουμε ούτε ένα εκατοστό από την εθνική μας ταυτότητα ή της γλώσσας μας αλλά ε, θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Είμαστε μία Ευρώπη αξιών ελευθερίας, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Ως λετονός μπορώ να πω ότι γνωρίζουμε τι σημαίνει να ζούμε ανελεύθεροι, χωρίς δημοκρατία και χωρίς κράτος δικαίου. Αυτό κανένας δεν χρειάζεται να το βιώσει ποτέ. έχουμε έναν ε, βασικό τρόπο για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Οικονομική Ένωση. Και είναι κάτι απλό. Καλύτερη η αγορά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλύσουμε τους φραγμούς της ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσουμε το περιβάλλον έτσι ώστε οι δικές μας εθνικές εταιρείες, ε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι επιτυχείς παίκτες στη διεθνή σκηνή. Αυτό είναι στο χέρι μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο θέμα του μεταναστευτικού ενισχύοντας ε, τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί όταν ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα μπορούμε να διατηρήσουμε ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα και να μην παρεμποδίσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μπορούμε να έχουμε μια ευφύ μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και πάλι το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις της αγοράς υπάρχουν και λειτουργούν. Αφήστε την αγορά να απορριθμίσει τις ενέργειες και η πράσινη ενέργεια θα απογειωθεί, θα απογειωθούν οι ευφύς τεχνολογικές λύσεις, θα συμμετέχουν οι καταναλωτέ και η αγορά θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Και σε ό,τι αφορά την κοινή μας ασφάλεια. Δεν βλέπω αντίφαση μεταξύ του να συμμετέχει κανείς στο ΝΑΤΟ όπως η χώρα μου και ισχυρότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέλος της ε, Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά θα πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από τη στρατιωτική ασφάλεια. Μιλάμε για την ε, ασφάλεια των πληροφοριών στο περιβάλλον πληροφοριών όπου ζουν οι πολίτες και θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την εκπόνηση νομοθεσίας προκειμένου να δούμε ποια είναι η ευθύνη των πλατφορμών ε, κοινωνικής δικτύωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ε, γιατί πολλές φορές η δράση τους παρεμποδίζει τη δημοκρατική ανάπτυξη. Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται απαραίτητα να πολεμήσουμε τους λαϊκιστές. Οι πολίτες ακούν τους λαϊκιστές γιατί είναι δυσαρεστημένοι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τις βασικές αιτίες. Ως Ένωση είμαστε πιο ισχυροί, όπως το δεμάτι από τις βέργες. Παίρνεις μια βέργα και σπάει. Ένα, ένα έθνος μας μπορεί να σπάσει όλα τα έθνη παγκοσμίω είναι μικρά, αλλά ενωμένοι είμαστε σαν αυτό το δεμάτι από τι Βέργες που δεν μπορεί να σπάσει και μπορούμε τη δική μα ιδέα του ελεύθερου αγοριού και του ε, εμπορίου και του τρόπου ζωή μπορούμε να την προωθήσουμε στι άλλε αγορέ και όχι να αφήσουμε του άλλου να επιβληθούν σε εμά. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη που είναι της ε, αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, μαζί με τις αξίες της ενέας αγοράς, να τις προωθήσουμε, να το κάνουμε αυτό με έναν ειρηνικό τρόπο, μέσω του διαλόγου, μέσω της συμμετοχής των πολιτών και έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά σας. Ευχαριστώ πολύ.